στις 13 ε, Σεπτεμβρίου 2012. Τα συνοπτικά πρακτικά και τα κείμενα που εγκρίθηκαν στις 13 Σεπτεμβρίου είναι στη διάθεσή σας. Έχετε αντιρρήσεις σε ό,τι αφορά τα συνοπτικά πρακτικά. Όχι. Ο κύριος Μπάρι Μάτλενερ μου ε, γνωστοποίησε την παρέτησή του από μέλος του Ευρωπαϊκού